I think that we could start. Please use your headphones because I will speak in my mother language. Θα μιλήσω στα ελληνικά, στη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ ε, για την ε, παρουσία σας εδώ. Είναι αρκετά νωρίς για μια συνέντευξη τύπου. Ε, λέγομαι Δημήτρης Παπαδημούλης, είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και είμαι και μέλος του Steering Committee μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μιας καινούρια συμμαχίας που λέγεται Progressive Caucus. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η πρωτοβουλία, είναι ένα φόρουμ διαλόγου και κοινή δράσης που συγκεντρώνει ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, την Ευρωομάδα της Αστεράς, την οποία Προσωπικά ανήκω, όπως και το κόμμα μου, την ομάδα των Πρασίνων και την Σοσιαλιστική Ομάδα. Είμαστε ευρωβουλευτές που παρά το ότι μας ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, έχουμε κοινέ ανησυχίες, κοινούς προβληματισμούς και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το φόρουμ για να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ανοίξουμε ένα διάλογο σε θέματα εξαιρετικά επίγοντα, για το πού πάει η Ευρώπη, τι θέλουν από την Ευρώπη οι πολίτες και τι δεν βρίσκουν από τις κυρίαρχες πολιτικές και για να αντιπαραταχθούμε και στην ατζέντα της λαϊκίστικης άκρας δεξιάς που επωφελείται από την κρίση της υπαρκτής Ευρώπης για να προτείνει τη δική της επιστροφή σε ένα άγριο και επικίνδυνο παρελθόν. Αλλά εκτός από τη συζήτηση αποφασίσαμε στα θέματα που μας ενώνουν κοινέ ανησυχίες και κοινοί προβληματισμοί να οργανώνουμε και κοινέ δράσεις. Μια τέτοια πρώτη κοινή δράση είναι η σημερινή πρωτοβουλία που οργανώνουμε για να συζητήσουμε με τη βοήθεια ειδικών και προσωπικότητων με σημαντικό κύρος τις συνθήκες της ΣΥΤΑ και της TTIP που θεωρούμε ότι φέρουν πολλούς κινδύνους για τα standards των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων. Ε, φιλοδοξούμε να έχουμε συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε ενημερώσει και τις ηγεσίες των τριών πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκουμε ότι δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική ομάδα, αλλά προσπαθούμε να ενισχύσουμε ένα διάλογο και κοινέ πρωτοβουλίε ανάμεσα στι προοδευτικέ δυνάμει του φάσματο του Ευρωκοινοβουλίου, που νομίζω ότι είναι επίγον και χρήσιμο για όλου. Πριν δώσω το λόγο στου συναδέλφου μου που θα μιλήσουν γι' αυτό, και να είμαι πάρα πολύ σύντομο, να σας πω ότι στις μέχρι τώρα συναντήσεις που έχουμε οργανώσει εσωτερικού διαλόγου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν συμμετάσχει περίπου 100 ευρωβουλευτές από τις τρεις πολιτικές ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή μας η πρωτοβουλία έρχεται να ανταποκριθεί σε μια υπαρκτή ανάγκη. Θέλουμε και τη δική σας συμβολή και με την παρουσία σας στην σημερινή μας συζήτηση, αλλά και θα σας κρατούμε ενήμερος για τη συνέχεια των πρωτοβουλειών μας. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον επόμενο συνάδελφο, τον Κιγιόν Μπάλας. Yes, I'm, uh, speaking in French. Uh, Θα μιλήσω γαλλικά. Λέγομαι Κιγιόν Μπάλας, ή μεγάλος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής από την περιοχή του Παρισιού, από το Ile de France. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία μονάχα σε αυτά που είπε ο Δημήτρης. Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω ότι ο χώρος αυτός που δημιουργούμε για συζήτηση μεταξύ προοδευτικών βουλευτών είναι ένας χώρος ανοιχτός, ο καθένας μπορεί να έρθει με τους δικούς του στόχους που μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά είναι και συμπληρωματικοί. Είναι ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων και κοινή δράσης. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για συμφωνίες όπως η ΣΕΤΑ. Συγχρόνως όμως, προωθούμε μια ιδέα που είναι ευρύτερη ότι σήμερα η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη απαιτεί μια πολιτική ανασύνθεση κατά κάποιο τρόπο όπου η αριστερά ή οι αριστερές δυνάμεις θα πρέπει να προετοιμάσουν μια τέτοια αλλαγή μέσα στην Ευρώπη. Είναι βέβαια φυσιολογικό κάποιοι να είναι πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με ένα τέτοιο στόχο από άλλους, αλλά η ανάγκη να υπάρξει μια προοδευτική συμμαχία μέσα στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφής. Είναι απαραίτητο να βρεθούμε σε ένα πιο στρατηγικό χώρο σε ό,τι αφορά τη δράση της αριστεράς τα επόμενα χρόνια μέσα στην Ευρώπη. Και το θέμα της συμφωνίας ΣΕΤΑ αυτή τη στιγμή. Ε, εκπληρεί περίπου δύο στόχους αν θέλετε, γιατί πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι παντού στον κόσμο υπάρχει μια φάση παγκοσμιοποίησης η οποία φτάνει στο τέλος της. Υπήρξε αυτή η ουτοπία μιας ευτυχισμένης παγκοσμιοποίησης που θα βασιζόταν στην ελεύθερη συναλλαγή <clears throat> εμπορευμάτων και υπηρεσιών και στη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς. Είδαμε τώρα ποιε είναι οι καταστροφικέ συνέπειε σε οικονομικό επίπεδο, φυσικά ακόμα περισσότερο σε κοινωνικό επίπεδο με όλο μεγαλύτερε ασυμμετρίε και ακόμα και σε δημοκρατικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι οι λαοί θέλουν να ξαναπάρουν στα χέρια την τύχη του και αυτό είναι πάρα πολύ φανερό και αυτό φαίνεται και σε συμφωνίες όπως η συζήτηση για τις συμφωνίες όπως η ΣΕΤΑ και η TTIP. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά αυτή είναι κάπως στο περιθώριο, κανείς δεν μιλάει για αυτήν. Αρκεί όμως να δει κανείς τι σημαίνει αυτή η συμφωνία στον τομέα της ενέργειας και επομένως η συνέπεια σε οικολογικό επίπεδο με την ε, διαπερατότητα των ε, ενεργειακών προϊόντων από τη μια πλευρά και την άλλη, όπου δεν θα υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές του περιβάλλοντος και με κινδύνους για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική καμπή. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία την ΣΕΤΑ πριν από την έγκρισή τη, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έχει υπάρξει εντελεχή ανάλυση τη. Η ΣΕΤΑ σήμερα και η συζήτηση γύρω από τη ΣΕΤΑ θα επιτρέψει στι προοδευτικέ δυνάμει να συνενωθούν, τουλάχιστον να έχουν μια κοινή αναγνωσή του κειμένου αυτή τη συμφωνία και να κατέβουν σε ένα αγώνα εναντίον τη, εάν το θεωρήσουν απαραίτητο. Δίνω το λόγο στην Εύα Ζολή, Ευρωβουλευτή των Πρασίνων. Καλημέρα. Ο, το προοδευτικό αυτό φόρουμ είναι για μας απαραίτητο ως η αναζήτηση και ενός τρίτου δρόμου για να ξεπεράσουμε τον μεγάλο συνασπισμό που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό χώρο για να συζητήσουμε τις δικές μας θέσεις και να αντιμετωπίσουμε κέρια θέματα όπως είναι η Συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και με τις επιτροπές έρευνας όπου θα πρέπει να δράσουμε από κοινού για να διαμορφώσουμε ένα πολιτικό χώρο ο μπορεί να αρθρώσει εναλλακτικέ θέσεις και όπως κάναμε στις επιτροπές έρευνας TAX 1 και 2 για τα φορολογικά θέματα θέλουμε να προωθήσουμε αυτή τη δημιουργία του εναλλακτικού χώρου και σε άλλους τομείς για να καταδείξουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει ένας χώρος που ανήκει στους πολίτες ώστε να μπορούν να προωθήσουν τη θέση τους και τη θέλησή τους στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να είμαι εδώ μαζί σας και μπορώ να συμβάλλω στην παρουσίαση αυτού του εγχειρήματό μας που είναι ακόμα σε ένα εμβριακό στάδιο όπως βλέπετε. Ελάτε λοιπόν σήμερα το βράδυ να ακούσετε τις αναλύσεις που θα παρουσιαστούν για τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, μια συμφωνία που προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν ουσιαστικά παρακάμπτοντας ακόμα και την διαβούλευση με, τον, το Κοινοβούλιο είναι απαραίτητο να γίνει μια ανάλυση προς όφελος και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κατανοήσουμε όλοι τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή και ιδίως για τους Γάλλους Γεώργους. Όλα αυτά λοιπόν έχουν παρασιοποιηθεί και γι' αυτό είναι απαραίτητο οι προοδευτικές δυνάμεις να συνενωθούν για να κάνουν ανάγλυφες όλες τις συνέπειες οι οποίες μπορούν να προκύψουν από αυτήν την συμφωνία. Είναι μια συμφωνία για την οποία δεν έχει γίνει καν μια <clears throat> έκθεση, μια ανάλυση αντικτύπου για τα αποτελέσματά της. Είναι η συμφωνία λοιπόν η οποία είναι πρόγευση της ταύτα μιας συμφωνίας με την ε, ε, Αμερικανική Ήπειρο και επομένως είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλύσουμε για να δούμε τι κινδυνεύουμε να έχουμε στο μέλλον. Ο Φάμπιο Τεμάση τώρα από την QNG έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Um, good morning to Καλημέρα σε όλους σας. Ε, είμαι ο Φάβιο Ντεμάση, ε, είμαι στην, Επιτροπή, στην Ερευνητική Επιτροπή για τα ε, Panama Papers μαζί με την ΕΒΑ και τον Πρόεδρο, αλλά τώρα μιλάω εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό μου. Έχουν περάσει λοιπόν διακοπές και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλήσω γερμανικά. Αυτός ο προδεκτικός πυρήνας είναι μια ε, πρωτοβουλία, ε, μια I think that there is German translation, am I correct? Yeah. Okay, it's good. Okay. Wir haben uns zusammengefunden, auch bei unterschiedlichen... Λοιπόν, Έχουμε σίγουρα διαφορετική παράδοση, αλλά αποφασίσαμε να συνεργαστούμε γιατί όλοι μας συμφωνούμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μια ολέτρια πολιτική στην Ευρώπη. Δεν με ακούτε. Είμαστε στο 7. Στο 7 είμαστε, είναι εντάξει. Στο 7. Και με ακούτε τώρα, εντάξει. Έχουμε λοιπόν ε, πολλές κρίσεις που βιώνουμε, την προσφυγική κρίση, το Brexit και πάρα πολλά άλλα, ε, κρίση οι οποίε ε, θα μας πλήξουν ουσιαστικά αν δεν ε, αντιδράσουμε. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζούμε μια, ένα είδος μεγάλου συνασπισμού και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις απλά και μόνο με τον αδρανή. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσει και πρέπει να κινητοποιηθούν οι ευρωβουλευτές. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι και στη Γερμανία στην σοσιαλδημοκρατία υπάρχουν ε, πλέον συζητήσεις ε, για, ε, το, για τη συμφωνία ΣΕΤΑ και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι στην πολιτική μας ομάδα, σε εμά στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις και υπάρχουν και πάρα πολλές επιφυλάξεις γενικότερα στους Γερμανούς πολίτες και αυτό είναι πάρα πολύ καλό το ότι συνδικάτα, φιλανθρωπικοί οργανισμοί, ακόμα και εκκλησιαστικοί οργανισμοί αντιδρούν έναντι αυτής της συμφωνίας. Ε, εμείς δεν πιστεύουμε όλα αυτά που μας υπόσχονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Και ο κύριος Ολόντ και ο κύριος Γκάμπριελ στη Γερμανία λένε πέθανε ε, το TTIP. Όμως υπάρχει η ΣΕΤΑ. Η συμφωνία ΣΕΤΑ είναι ο μικρός αδελφός, η μικρή αδελφή αν θέλετε τη συμφωνία TTIP. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι Γερμανοί ε, δικαστές τοποθετήθηκαν και είπαν ότι οι επιχειρήσεις αν τα κράτη παρεμποδίζουν τον προσπορισμό κερδών, δίνονται να καταφύγουν σε αυτά, στα δικαστήρια. Υπάρχει αυτό, αποφασίστηκε στη Γερμανία. Εμείς θα εξετάσουμε και άλλα επίμαχα θέματα επί των οποίων θα συζητάμε με τους ευρωβουλευτές. Όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Παπαντιμούλης, ε, υπάρχουν 50, άλλες φορές 100 άνθρωποι που συζητούν ε, με διαφορετικές απόψεις, αλλά σε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα, γιατί ξέρετε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε αρκετό καιρό για να μπαίνουμε στην ουσία των θεμάτων, σε πολιτικές ουσιαστικές συζητήσεις. Εμείς ε, θέλουμε να συμμετάσχουμε και σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο των εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί θέλουμε να συσφίξουμε τους, ε, θεσμούς, τους ε, δεσμούς μας ε, με τους, με τους Βρετανούς εργατικούς. Δεν θα σας ενημερώσουμε σήμερα για όλα μας τα σχέδια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε τα προγράμματά μας. Ευχαριστώ. Oh, έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ο κύριος Ουρτασούν από τους Πράσινους και μετά θα έχουμε περιορισμένο χρόνο για συζήτηση. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά επίσης, ώστε να καλύψουμε όλο το φάσμα γλωσσών σήμερα εδώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Εν συντομία, μερικές σκέψεις θέλω να σας αναφέρω. Πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε συνεργαστεί ήδη στο παρελθόν για τη δημιουργία αυτής της ομάδος και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με την ε, ε, συνέντευξη τύπου τώρα και με την απογευματινή εκδήλωση ξεκινούμε τις δραστηριότητές μας και επισήμως, θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πραγματικό κενό. Εγώ ένιωσα μεγάλη ε, έκπληξη γιατί είδα ότι δεν υπήρχε κάποιος χώρος συζήτηση μεταξύ των δυνάμεων της αριστεράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Όλοι μας έχουμε ε, αποδηθεί σε αγώνες με, με απόψεις πολύ κοντά ημέν των δε, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ένα κοινό χώρο, ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε με αυτό το προοδευτικό χώρο, το προοδευτικό φόρουμ το οποίο δημιουργούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία γιατί πρέπει να μην κρατήσουμε τις σκέψεις μας, τις κριτικές μόνο στον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να τις ανταλλάξουμε μεταξύ μας για να έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε. Βρισκόμαστε όμως και σε ένα, ένα δεύτερο κενό που έχει ακόμα μεγαλύτερο, μεγαλύτερη διάσταση και αφορά όλη την Ευρώπη, ότι οι πολίτες της Ευρώπης δεν έχουν μπροστά τους κάποιες σαφείς ιδέες της αριστεράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα κενό σε σχέση με τις προτάσεις της ε, αριστερής σκέψης. Έχουμε μια χρονική στιγμή γεμάτη προβλήματα και δυσκολίες. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να γεμίσουμε αυτό το κενό με προτάσεις δικές μας και να δημιουργήσουμε ένα τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα με διάλογο, με φόρου, με κοινά βήματα συζήτησης Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και θα ήθελα να κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση και ερω... ερωτήσεις και σύντομες ε, απαντήσεις. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ε, Πασκάλ Βερντό από την Φαστιβιζιό για την ε, ΣΕΤΑ κυρία Ζολή, αν θέλετε να απαντήσετε. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέπει την ε, ε, εισαγωγή βοήου κρέατος, περίπου 500.000 τόνους και εσείς καταγγέλλετε την έλλειψη διαφάνειας έναντι των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνομοσπονδία των παραγωγών βοήου κρέατος η οποία έχει κάνει μια στη Γαλλία και κάπως έχει παρακαμφθεί η προσπάθειά τους. Σημερίζεστε την ε, τις ε, ανησυχίες τους σε σχέση με την εξαφάνιση ορισμένων είδων, ειδών βοηδών όπως είναι τα σαρολέ στη Γαλλία. Και επίσης λένε πολλοί ότι πολλά από αυτά τα, βόια, τα προϊόντα βόηου κρέατος από τον Καναδά θα είναι γεμάτα ορμόνες. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Και εγώ συμμερίζομαι απόλυτα αυτές τις ανησυχίες, τις ανησυχίες των παραγωγών βοήου κρέατος στη Γαλλία 60.000 τόνοι ε, βοήου κρέατος, ακόμα και αν υψηλής ποιότητας θα διαταράξουν την αγορά και εξάλλου αυτή τη στιγμή 40% των ε, εξαγωγών από βοήου κρέατος από τον Καναδά πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Και Τώρα αυτή η ποσότητα θα πρέπει να περάσει στις υπόλοιπες 27 χώρες άμα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο στόχος αυτής της συμφωνίας, ο δεδηλωμένος στόχος, είναι να ξεπεραστούν όχι μονάχα τα τελωνιακά εμπόδια που δεν υπάρχουν πια ουσιαστικά, αλλά και τα φυτογειονομικά πρότυπα να ξεπεραστούν που είναι κέρια για τη δημόσια υγεία και όπως είπατε και για τη διατήρηση των ηθαγενών ζωικών ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση και να βοηθήσουμε τους πολίτες της Ευρώπης να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Και επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή τη συνθήκη, για να μπορέσει να την απορρίψει πρέπει να υπάρχει πίεση της κοινή γνώμης. Αυτός λοιπόν και είναι ένας, και είναι και ένας τρόπος να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που μας αφορά όλους και το οποίο προσπαθούν πολλοί να περάσουν στα μουλοχτά χωρίς να υπάρχει γνώση της κοινή γνώμης. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι στις ερωτήσεις αλλά και στις απαντήσεις, λέει ο κ. Παπαδημούλης. Καλημέρα σας. Ποιος είναι ο στόχος της εκστατείας σας. Τι θέλετε να επιτύχετε. Θέλετε να υπάρξει διαπραγμάτευση της συμφωνίας ΣΕΤΑ. Να υπάρξει κάποια άλλη ενέργεια σε σχέση με τα θέματα αυτά. Και δεύτερον, και το δεύτερο ερώτημά μου είναι αν σκέφτεστε για τη συμφωνία με το, εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ με τη Σιγκαπούρη που πλησιάζουν το στάδιο της οριστικοποίησης τους από τις συμφωνίες. Και τέλος για την πλατφόρμα σας. Λέτε ότι είσαστε ένας χώρος πολιτικής ε, προβληματικής και συζήτησης, ένα κόκκους όπως λένε, αλλά συγχρόνως είσαστε κατά τη ΣΕΤΑ που θεωρείται μια από τις πιο προοδευτικές ε, συμφωνίες σε εμπορικό επίπεδο. Πώς, τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά λοιπόν. Πάρα πολύ σύντομα, εγώ θα μιλήσω μόνο εξ ονόματός μου, αλλά νομίζω ότι και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορούμε να κυρώσουμε τη συμφωνία ΣΥΤΑ ως έχει. Ε, μας ενδιαφέρει να την ε, παρεμποδίσουμε, την εφαρμογή της ε, και σε προκατρακτική φάση πάρα πολλά κράτη-μέλη, τελικά ε, κυρωθεί αυτή η συμφωνία, πάρα πολλά κράτη θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ε, υπάρχει και πρόβλημα για το κατά πόσον θα περάσει από τα κοινοβούλια αυτή η συμφωνία. Όχι, συμφωνώ με το αυτό που είπατε για τον πυρήνα μας, για τον κόκκους, ότι είναι προοδευτικός. Αλλά αν θέλετε θα μας επιτρέψετε να επανέλθουμε σήμερα το απόγευμα που θα το εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Εμείς ε, δεν είμαστε ομάδα πίεσης για εμπορικά θέματα. Εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα, στο, στη μετανάστευση, στο dumping στην ανάγκη επενδυτικών προγραμμάτων. Αλλά μέχρι τώρα, και αν θέλετε μπορείτε ε, να πάτε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ήδη από τη σύσταση κοινής αγοράς μας είχαν υποσχεθεί ανάπτυξη και απασχόληση και αυτά δεν έγιναν. Έχουμε λοιπόν ε, πολλές ε, ενδείξεις ε, για το ότι σήμερα πλέον υπάρχει ουσιαστική κρίση της δημοκρατίας στις εκλογές προχτές στη Γερμανία, είδατε τι έγινε με τους ακροδεξιούς, οφείλουμε να τοποθετηθούμε έναντι αυτού. Είμαι από την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Ε, μερικοί από εσά αναφερθήκατε στο μεγάλο συνασπισμό που υπάρχει στο Κοινοβούλιο και θέλω να ρωτήσω, στόχο έχετε να επιτεθείτε σε αυτό το μεγάλο συνασπισμό έτσι ώστε να διαλυθεί ενδεχομένως αυτό ο συνασπισμός ε, και επειδή άρχισα λιγάκι να μην το πρόλαβα, ε, μήπως μπορείτε να μα πείτε τα μέλη, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το κόκκου. Κυρίω μπορείτε να μου πείτε αν θα υπάρχει κάποιο από του Γερμανού Σοσιαλδημοκράτε, από το S5 που θα συμμετέχει σε αυτό τον ε, Για το θέμα του βοήου κρέατος, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως, θέλω να τονίσω πόσο παράλογο είναι να διακινείται βόλιο κρέας σε παγκόσμιο επίπεδο τη στιγμή που μπορούμε να παράγουμε τέτοια προϊόντα σε τοπικό επίπεδο. Και επομένως αυτό θα είναι μια άμεση προοδευτική συνέπεια αν δεν γίνει αυτή η συμφωνία και δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι είναι προοδευτική αυτή η συμφωνία πέραν αυτών οι οποίοι έχουν συμφέρον να περάσει αυτή η συμφωνία. Ένα δεύτερο στοιχείο, κάτι, πιο, κάτι ευρύτερο κάπως, ο στόχος σήμερα του προοδευτικού αυτού κόκκους, αυτού του, της ομάδος πολιτικής δράσης, είναι να αντιμετωπίσουμε γενικά το θέμα των ελευθέρων συναλλαγών. Δεν είμαστε κατά των διεθνών συναλλαγών δεν είμαστε προστατευτιστέ, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι διεθνεί εμπορικέ συναλλαγέ ανταποκρίνονται σε κοινωνικά, οικολογικά ε, πρότυπα τα οποία να είναι βιώσιμα και δεν έχουν μόνο γνώμονα το κέρδο. Επίση. για την δυναμική τη ομάδα μα. ναι, πράγματι υπάρχουν μέλη του s 5 που έρχονται τακτικά στι συνεδριάσει μα. Δεν είναι μέσα στην ε, κατευθυντήρια ομάδα που βρίσκεται εδώ στο ε, που βρίσκεται εδώ μπροστά σας, αλλά συμμερίζονται τις ε, επιθυμίες και τους στόχους μας για τον μεγάλο συνασπισμό. Η ιδέα μας δεν είναι να έχουμε μια τελείως διαφορετική στρατηγική μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δημιουργήσουμε προβλήματα στις πολιτικές ομάδες. Θέλουμε να δείξουμε όμως ότι υπάρχει αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τους σοσιαλιστές να δίνουν πάντα την ε, προτεραιότητα στην, στο συνασπισμό με τη δεξιά χωρίς να συζητήσει με τις άλλες αριστερές ομάδες. Ξέρω ότι εσείς ε, έχετε αυτές τις επικρίσεις για τη ΣΕΤΑ σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των επενδυτών. Σας ε, ενοχλεί η μορφή της ΕΤΑ είσαστε εναντίον γενικά των συμφωνιών ελευθερίου εμπορίου. Αν υπήρχαν συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, πώς θα τις διαμορφώνετε εσεί, πώς θα θέλατε να είναι αυτές οι συμφωνίες. Κοιτάξτε, η συζήτηση δεν είναι γενική φύση για το ελεύθερο εμπόριο. Εμά μα απασχολούν πολύ ε, συγκεκριμένα θέματα. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε πιο συγκεκριμένα θέματα, γιατί σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε ακριβώ αυτή την ανάγνωση των κειμένων και θα ε, καταλήξουμε ε, σε συγκεκριμένα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, μα απασχολούν, παραδείγματο χάρη, ο μηχανισμό διαιτησία. Αυτό μα απασχολεί. Είναι κάτι που μα απασχολεί Πολύ πολύ, είναι σαφές. Και όπως είπε και ο Γκυγιόμ, οι επιπτώσεις στην ε, γεωργία και κάποια άλλα συναφή θέματα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι σήμερα το απόγευμα δεν θα κάνουμε έτσι γενικές συζητήσεις ε, για το ελεύθερο εμπόριο, αλλά θα μπούμε σε λεπτομέρειες ε, του κειμένου. Και νομίζω όλοι σας γνωρίζετε ότι έχουμε συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με τα κείμενα. Eric Bonze από την ε, Tageszeitung και θέλω να κάνω μία ερώτηση για την άκρα δεξιά. Η άκρα δεξιά ισχυρίζεται ότι είναι κατά των συμφωνιών ΣΥΤΑ και ΤΙΤΙΠ. Τώρα εσείς αυτό πώς το αξιολογείτε. Σα δημιουργεί πρόβλημα ότι είναι και αυτοί κατά. Ε, όχι, δεν είναι πρόβλημα ε, το ότι ισχυρίζεται κάτι ακροδεξιά, γιατί ξέρετε γιατί, γιατί εμείς κάνουμε κάτι, δεν ισχυριζόμαστε απλώς, δεν παραμένουμε στα λόγια. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι αρκεί να διαμαρτύρεται κανείς για την άνοδο της ακροδεξιάς ε, στις χώρες μας, πρέπει να κάνουμε αναλύσεις. Πώς έγινε κάτι τέτοιο, από πού προέρχεται. Είναι οι αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές που είναι κατοχυρωμένες και σε συμφωνίες ε, όπως η ΣΥΤΑ ή παλαιότερα για την κοινή αγορά. Αν δείτε και την ε, ψηφοφορία, το δημοψήφισμα για το Brexit, εκεί θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένους φόβους. Κοινωνικό dumping, παραδείγματος χάρη. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα προστατεύοντας ε, τις συμφωνίες ε, συλλογικών ε, συμβάσεων και αυτό όμως δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι την ακροδεξιά μπορεί κανείς να την πολεμήσει κατά τον καλύτερο τρόπο αντιμετωπίζοντας τις αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος. Τώρα η ακροδεξιά ισχυρίζει ότι είναι κατά του TTIP και τη ΣΥΤΑ. Εγώ έχω δει πάρα πολλούς ακροδεξιούς ε, που συνυπέγραψαν ε, μαζί με το ε, μεγάλο συνασπισμό αυτές τις συμφωνίες. Οι αρχές της EFD, ο Μπέρντ Λούκε τότε που συμμετείχε και αυτός είχε υπογράψει. Όπως είπε ο Φάμπιο, η ατζέντα και οι στόχοι του Progressive Caucus είναι στον αντίποδα της λαϊκίστικης ακροδεξιάς. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη, ισχυρό κοινωνικό κράτος, ενίσχυση των πολιτικών συνοχής, ευρωπαϊκές λύσεις στο προσφυγικό, εφαρμογή των στόχων που προστατεύουν τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή, περισσότερη δημοκρατία και όχι επιστροφή σε ένα κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Και διαπιστώνουμε καθημερινά ότι πολλές φορές η ρητορική της άκρας δεξιάς εμφανίζει ορισμένους δήθεν κοινωνικούς στόχους, αλλά η ατζέντα τους είναι επιστροφή στο παρελθόν. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία που θέλει να ανοίξει πόρτες για το μέλλον. Ο στόχος μας δεν είναι να καταστρέψουμε άλλες συμμαχίες, αλλά να κάνουμε την Ευρώπη πιο ελκυστική για τους πολίτες της, πιο δημοκρατική, πιο κοινωνική, γιατί η σημερινή Ευρώπη δεν αρέσει και η αποτυχία των κυρίαρχων πολιτικών είναι αυτή που τρέφει την άκρα δεξιά. Άρα θα σας έλεγα ότι προσπαθούμε να διαμορφώσουμε με διάλογο, με σκληρή προσπάθεια, την τρίτη εναλλακτική λύση απέναντι στη σημερινή κρίση και απέναντι στην επιστροφή στο παρελθόν, το άγριο και το φοβικό παρελθόν που εκπροσωπεί η άκρα δεξιά. Δεν ακούγεται ο μιλητής δυστυχώς. Νομίζω ότι ο χρόνος μας τελείωσε. Σας προσκαλούμε να έρθετε στο, στην εκδήλωσή μας στις 6.30 το απόγευμα. Και ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς. Γιατί καταδαπανίσαμε 5 λεπτά παραπάνω από το προβλεπόμενο.